Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε την συνάντησή μας σήμερα καλωσορίζοντας τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μισελ Σαπέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου με σας και τη χώρα σας. είναι η πρώτη επαφή μετά από την εφαρμογή του εξαπλού πακέτου και η παρουσία σας εδώ εκτιμάται δεόντως. Όπως είδατε την προηγούμενη Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε στις προβλέψεις της ότι υπάρχει μια θετική τάση στη Γαλλία σε σχέση με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, όπως και με τις περισσότερες άλλες κοινοτικές χώρες και ο δρόμος της μείωσης των ελλημάτων είναι ένας δρόμος που αποδίδει περισσότερο από όσο υπολογίζαμε. Βλέπουμε τα αποτελέσματα για το 2014. 4%, 3,8% το 2015, ενώ παλιά λέγαμε για 4,3% και 4,1%. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για ευελιξία γενικότερα, αλλά σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για μια κάποια πρόοδο. Οι αριθμοί λοιπόν επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική η οποία ακολουθείται και η οποία έχει σαν στόχο να κατέβει το έλλειμμα κάτω από το 3% για τον επόμενο χρόνο. Συνεχίζεται επίσης και ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στον Υπουργό να ακούσουμε τις απόψεις του και για τη Γαλλία, αλλά ίσως και για άλλα θέματα ευρύτερα που αφορούν στην Ευρώπη, τις προβλέψεις για την Ευρώπη και θέματα μεταρρύθμισης στον κλάδο της οικονομικής διακυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Να πω σε όλους, όταν φορέσετε τα ακουστικά σας, να πω λοιπόν στον καθένα από σας ότι με χαρά σας συναντώ. Λέτε ότι είναι πρώτη φορά που η Γαλλία συμμετέχει σε αυτόν τον διαρθρωμένο διάλογο στα πλαίσια των νέων ρυθμίσεων. Χαίρομαι που είμαι εδώ πρώτος. Ε, περιμένετε τη Γαλλία και χαίρομαι που μας περιμένετε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε και εμείς παρόντες προετοιμασμένοι. Η συνάντηση αυτή είναι καλό που γίνεται. Ένα χρόνο μετά από την άνοδο στην, από, από τον σχηματισμό της νέας γαλλικής κυβέρνησης του κυρίου Βάλς και ένα χρόνο παρουσίας δικής μου στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ένα Υπουργείο που γνωρίζω γιατί είχα περάσει ήδη από το 92-93 πριν από το ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών στη Γαλλία. Είμαι άνθρωπος που έχω εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και ε, πιο συγκεκριμένα στον κλάδο μου της Οικονομικής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες ε, βασικές αρχές στην επικοινωνία μας. Ε, θα μπορέσετε να θέσετε λοιπόν τις ερωτήσεις σας και να δώσω απαντήσεις. Να μιλήσω λίγο για την κατάσταση όμως να μου επιτρέψετε στη Γαλλία. Και όταν θα μιλήσω για τη Γαλλία θα μιλήσω και για την Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν ε, τρομερές διαφορές ανάμεσα στην σφαιρική κατάσταση από τη μία και στην κατάσταση σε κάθε μία χώρα από την άλλη. Γνωρίζω ότι η Γαλλία ε, και εδώ και αλλού είναι θύμα διαφόρων έτσι κλισέ θα έλεγα και σε κάθε κλισέ βέβαια υπάρχει μια κάποια δόση αλήθειας. Είναι βέβαια κάτι το οποίο εξελίσσεται, μια κατάσταση συνεχώς εξελίσσεται και έτσι λοιπόν και τα πράγματα στη Γαλλία αλλάζουν και στον τομέα του των σοβαρών μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής σωστότερης οργάνωσης. Η Γαλλία είναι σε θέση να σεβαστεί τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις, ταυτίζεται με αυτές τις υποχρεώσεις. Η Γαλλία ήδη από το 2012 έχει αναλάβει να φέρει πέρας μια βαθιά μεταρρυθμιστική πολιτική Νομίζω ότι οι σωστές μεταρρυθμίσεις είναι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει αντικείμενο διαβούλευσης και είναι σε θέση να αλλάξουν την οικονομική και δημοσιονομική μας κατάσταση. Για τα θέματα τα δημοσιονομικά τώρα. Είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν υποθέτω σας παθιάζουν θα έλεγα και ασκήσατε κριτική στο παρελθόν επανειλημμένα εις βάρος της Γαλλίας. Το είπατε Πρόεδρε ότι το 2014 ε, η Γαλλία πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενε κανείς και στον τομέα της μείωσης των ελλημάτων και στον δημοσιονομικό τομέα. Αυτοί δηλαδή που θα είχαν θεμητά ερωτηματικά τον Οκτώβριο αν η Γαλλία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της για το 2014 μήπως έχει ε, φτάσει η φάση να περάσει σε ε, περίοδο κυρώσεων δημοσιονομικών εις βάρος της Γαλλίας. Όχι. Ε, τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων αρχών και οργανισμών δείχνουν ότι το 2014 σεβάστηκε η Γαλλία τις υποχρεώσεις της εκτός από το θέμα του ελλείμματος. Για το 15 και 16 συνεχίζουμε με τις νέες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο και εκεί αναφέρατε κάποιους αριθμούς. Οι τελευταίες προβλέψεις λένε 3,8% έλλειμμα, ονομαστικό δημόσιο έλλειμμα. Αυτός είναι ακριβώς και ο στόχος, το ποσοστό που έχουμε θέσει και εμείς μόνοι μας και που συμπεριλαμβάνεται στην ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2015. Το ίδιο ισχύει και για το 2016 και το 2017. Η Γαλλία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, θα κατέβει το 2017 κάτω από το 3%. Απαιτούνται προσπάθειες, απαιτούνται προσπάθειες ελέγχου των δημοσιονομικών δαπανών. Το 2014 πήγε καλύτερα όπως είπα, όχι γιατί συλλέξαμε περισσότερους φόρους, γιατί και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες η ανάπτυξη στη ζώνη ευρώ θα έλεγα ήταν αρκετά χαμηλή. Αλλά γιατί ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμεινο κάναμε τεράστιες προσπάθειες ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Έξι δις βγάλαμε και αυτό επηρέασε ε, τα αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στα πλαίσια αυτής της εξοικονόμησης πιστώσεων, στα πλαίσια του προϋπολογισμού, μια μεγάλη προσπάθεια αλλά και στοχευμένη προσπάθεια έτσι ώστε να μην θίξει την ανάπτυξη. Αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο τίθεται για όλους. Πώς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σοβαροί στα δημοσιονομικά, να μειώσουμε το έλλειμμα για να μην αυξήσουμε μακροπρόθεσμα το χρέος, ενθαρρύνοντας όμως κάτω από τις σημερινές συνθήκες, τη σημερινή συγκυρία, την τόσο εύθραυστη, μια οικονομική ανάπτυξη η οποία αρχίζει να ανεβαίνει αλλά με αργές ταχύτητες. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε έτσι ώστε η τάση αυτή να επιβεβαιωθεί, να γίνει πιο μόνιμη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, περισσότερο ίσως σε άλλες χώρες, θέματα όπως η απασχόληση. Η Γαλλία λοιπόν θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της στον τομέα της σοβαρής αντιμετώπισης των δημοσιονομικών. Το δεύτερο κλισέ είναι αν γίνονται μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία. Φυσικά και γίνονται. Από το 2012 μεταρρυθμίζεται σε πάρα πολλούς τομείς η χώρα μου. Πρώτον, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ε, φύγεται η ανταγωνιστικότητα λόγω των ε, συνεισφορών, λόγω του κόστους γενικά του οικονομικού που επιβάλλεται από το κράτος. Εμείς διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα σε τέσσερα χρόνια που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 40 δις επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό πολλές γαλλικές επιχειρήσεις έχουν ισορροπήσει καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το 2010 και αυτό φαίνεται και στις προθέσεις τις επενδυτικές. Χτες είδαμε ότι υπάρχουν προθέσεις επενδύσεων συν 7% για το 2015 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο γιατί η ανάπτυξη τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τροφοδοτείται από τις εξαγωγές, αλλά λείπουν οι επενδύσεις, ιδιαίτερα οι ιδιωτικές επενδύσεις. Και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση και με τους στόχους της Νέας Επιτροπής και του Κοινοβουλίου φυσικά, πρέπει να ενθαρρυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα στις χώρες που έχουν ανάγκη. Δεύτερη πλευρά είναι αυτή η οποία αφορά την αγορά εργασίας, έτσι το λέμε. Ήμουν υπουργό Εργασίας πριν γίνω υπουργό Οικονομικών. Ασχοληθήκαμε και με το θέμα των συλλογικών ε, απολύσεων. Πρέπει να συνοδεύουμε σωστότερα και καλύτερα τους απολυμένους εργαζομένους. Θα πρέπει όμως να μην δημιουργούμε και εμπόδια στις επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν νέους ε, υπαλλήλους και θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας πάνω σε αυτά τα θέματα καλύτερα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πάντως η Γαλλία προχωρά και στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές δεν είναι βίαιες, είναι σταδιακές, είναι προοδευτικές, είναι καρπός διαπραγμάτευσης. Επιζητούμε την ευημερία, επιζητούμε όμως ε, ε, την ε, βιωσιμότητα αυτών Βλέπετε ότι παλιά λέγαμε ότι στη Γαλλία γίνονται συνεχώς απεργίες, υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές. Αυτά έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, έχω λίγα λεπτά ακόμα να μιλήσω λίγο όχι μόνο για την ε, Γαλλία αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε το 20%, 21% σε επίπεδο ΑΕΠ για το σύνολο της Ευρωζώνης. Έχουμε φίνες ως προς αυτό. Αλλά παρόλα αυτά ε, προσπαθούμε να χτίσουμε και την αυριανή Ευρώπη. Και θα ήθελα να αναφερθώ στις κοινέ προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρώτη προσπάθεια, το θέμα της φορολογίας. Δεν χρειάζεται να σας πω εδώ γιατί είναι κάτι το οποίο συμμερίζεστε. Το πόσο σημαντικό είναι να συγκλίνει κανείς τον τομέα των αγορών, να συγκλίνει σε επίπεδο πιστοτικών ιδρυμάτων, να συγκλίνει σε τομείς υπολογισμού του κόστους παραγωγής και του κόστους εργασίας, όταν από την άλλη έχουμε διαφορές, σημαντικότατες διαφορές για να μην μπορείξεις από τη μία χώρα στην άλλη σε επίπεδο φορολογικό. Χωρίς να προχωρήσουμε σε μια πλήρη φορολογική εναρμόνιση βέβαια στην παρούσα φάση, αλλά να θέσουμε τέλος σε ανώμαλες καταστάσεις φορολογικού ανταγωνισμού είναι μια ευθύνη για τη Γαλλία και έχουμε ε, ξεκινήσει μια πρωτοβουλία πρόσφατα με την Ιταλία και τη Γερμανία θα κάνουμε προτάσεις διαφανείς προτάσεις και για τα λεγόμενα tax rulings, τις ειδικέ φορολογικές ρυθμίσεις και να αποτρέψουμε την ύπαρξη μηχανισμών μεταφοράς κερδών αξίας που δημιουργείται σε διάφορες χώρες από τη μία χώρα στην άλλη για φορολογικούς λόγους. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν πολύ. Βλέπω πως πήγαιναν τα πράγματα πριν μερικά χρόνια. Ήταν αδύνατο, ήταν ασύλληπτο θα έλεγα, να θέλει κανείς να τερματίσει τέτοιες καταστάσεις. Σήμερα όμως είναι μια εκπεφρασμένη ανησυχία μας και πρέπει να προχωρήσουμε. Μια τελευταία λέξη και θα τελειώσω εδώ έτσι ώστε να υπάρξουν και ερωτήσεις όποιοι επιθυμούν. Σε αυτή την προσπάθεια διαβούλευσης, διαλόγου που ονομάζουμε Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι μια προσπάθεια χρήσιμη, είναι μια προσπάθεια απαραίτητη. Απαιτείται να λειτουργούμε με ευρωπαϊκό τρόπο, να σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και των διαφθορτικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη. Αυτή η σφαιρική αντίληψη θα πρέπει να προηγείται της εφαρμογής αναχώρα αν θέλετε αυτών των πολιτικών. Στο παρελθόν γιατί ήταν απαραίτητο ίσως, γιατί ήταν κατεπήγον ίσως λόγω ειδικών δυσκολιών αλλά υπήρχαν γενικά πολλές συνταγές και σκέψεις για το τι θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά και όχι για το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη συνολικά. Πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουμε τη μεθοδολογία μας. Είναι αυτό απαραίτητο. Τι θέλουμε σε δημοσιονομικό επίπεδο για την Ευρωζώνη. Και αφού το αποφασίσουμε αυτό, πώς θα εφαρμόσουμε αυτή την κοινή μας βούληση σε κάθε χώρα. Γιατί φυσικά κάθε χώρα είναι διαφορετική. Και οι μεταρρυθμίσεις, οι διαφορετικές που θα πρέπει να γίνουν σε κάθε χώρα θα πρέπει να γίνουν με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό χρονισμό. Αυτό θα μετριάσει τις συνέπειες και σε κοινωνικό επίπεδο και στον τομέα ε, των αγορών γενικότερα και στις υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά να δώσουμε συστάσεις σε κάθε χώρα, γιατί κάθε χώρα έχει ειδικέ ανάγκες, ειδικέ συγκυρίες κτλ. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να το κάνουμε και η Γαλλία θα προσπαθήσει έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα νοοτροπία, μια νέα αντίληψη σφαιρικής πρώτα επεξεργασίας θέσεων και μετά εφαρμογής αναχώρα, κάτι το οποίο θα είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε Ο μιλητές, ο κύριος Μπάλτς, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποφασιστικότητά σας και το θάρρος σας μεταξύ του οποίου και το γεγονός ότι ήρθατε ενώπιον της Επιτροπής μας. Και υπάρχει και ένα κοινό χρονοδιάγραμμα το οποίο αφορά αυτά που είπατε. Θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν στην αρχή της παρέμβασής σας ήδη αναφερθήκατε στο θέμα του ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γαλλίας. Το Σύμφωνο Σταθερότητος και Ανάπτυξης δίνει ένα, μια προθεσμία για να φτάσει κανείς σε εξισορροπημένο προϋπολογισμό. με μείωση κατά 2-3% κάθε χρόνο χρειάζεται να υπάρξει η κίνηση προς να φτάσει κανείς σε ένα προϋπολογισμό που θα φτάσει με έλλειμμα κάτω από το 3%. Η Γαλλία όμως ήταν τα τελευταία χρόνια με ελλείμματα του 3-3,5% του προϋπολογισμού της, ως αποτέλεσμα αυξάνεται η συνολική χρέωση της Γαλλίας και θα είναι σύντομα 100% του ΑΕΠ. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι το εξής. Με ποιο τρόπο θέλετε εσείς να επανέλθετε στα όρια τα οποία προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δηλαδή το 60% σε συνολικό κρατικό χρέος, ποια είναι τα χρονοδιγράμματά σας και τα μέτρα τα οποία θέλει να λάβει η κυβέρνησή σα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημά μου. Το δεύτερο θέμα είναι το κόστος του συνταξιοδοτικού. 14% του ΑΕΠ σα πηγαίνει αυτή τη στιγμή σε συντάξει. Υπάρχει εδώ μια σταθερή αύξηση του ποσοστού αυτού. Άλλες χώρες στην Ευρωζώνη και εκτός της Ευρωζώνης έχουν τα τελευταία χρόνια κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση. το να υπάρχει η ηλικία συνταξιδότηση 61 ετών, αυτό είναι από τις χαμηλότερες στις χώρες του ΟΣΑ. Γι' αυτό θα να σας ρωτήσω ποια είναι τα σχέδια τα οποία έχετε εδώ για να αναστρέψετε αυτή την τάση, η οποία βέβαια επέχει πολλούς κινδύνους για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαπέν. Δεν χρειάζεται μεγάλο θάρρος για να έρθω εδώ ενώπιον σας. Είναι χαρά αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ακόμα και να χρειάζεται να είμαι υπόλογος ε, και να λογοδοτήσω για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζω με θετικό πνεύμα. Εν συντομία λοιπόν, η Γαλλία ξεκινάει από πολύ μακριά σε ό,τι αφορά το έλλειμμα του προπολογισμού. Και η Γερμανία έχει ξεκινήσει από μακριά και χρειάστηκε και αυτή να περάσει ένα δρόμο δύσκολο, ίσως με πιο γρήγορα βήματα. Εμείς ήμασταν σε μια πιο δύσκολη κατάσταση πριν και από την κρίση του 2008, πριν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να κάνουν τις απαραίτητες ε, ενέργειες περιστολής των ε, ελλημάτων. Εμείς είχαμε όμως ένα συσσωρευμένο έλλειμμα από το παρελθόν, συν το αποτέλεσμα της κρίσης. Ξεκινάμε λοιπόν από πιο δυσμενή θέση και φυσικά είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα η οποία είναι μεγάλη να μπορέσουν να αλλάξουν εκ βάθρων τα, τις δομές τους και τις κοινωνίες τους. Το κάνουμε όμως αυτό. Η πρώτη μας προτεραιότητα η πρώτη απέτηση φυσικά είναι να μπορέσουμε να σεβαστούμε τις προοπτικές που έχουμε ήδη οι ίδιοι θεσπίσει μας με την Κομισιόν σε ό,τι αφορά το ονομαστικό έλλειμμα. Αυτό είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει επιτευχθεί αυτό πλήρως. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε αυτή τη φορά να το πετύχουμε. Το 3% ως όριο του ελλείμματος 2017 είναι εφικτό. Δεύτερον, μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο δεν πρέπει μέσα στα πλαίσια των ε, κανόνων του προπολογισμού που είναι θεμητοί, δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα τα οποία θα είναι τόσο αυστηρά ώστε θα σταματήσουν την μικρή οικονομική ανάπτυξη η οποία δημιουργείται και την οποία θέλουμε να την εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί. Στη δύσκολη αυτή στιγμή ανάκαμψη οικονομικής δραστηριότητας, η ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της προοπτικής μείωσης του ελλείμματος θα πρέπει να συνάδει με την προοπτική να διατηρήσουμε την ε, ε, οικονομική ανάκαμψη που απαιτεί και κάποια βοήθεια από τα κρατικά κονδύλια, από το κρατικό προπολογισμό σε αναπτυξιακό επίπεδο. Σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια σταθεροποίηση του δημοσίου χρέου κάτω από το 100% δεν θα φτάσουμε τελικά το 100% και φυσικά στη συνέχεια θα πρέπει να το μειώσουμε προς τους στόχους του μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως το οποίο τίθεται για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη Γερμανία ακόμα. Για το δεύτερο ερώτημά σας, πρώτα απ' όλα. Εμείς ξεκινήσαμε μια μεταρρύθμιση για τα θέματα των συντάξεων. Γίνεται σταδιακά φυσικά αυτή η μεταρρύθμιση. Η ηλικία της ε, συνταξιοδότησης σταδιακά ανέρχεται λέτε είναι 61 η ηλικία συνταξιοδότηση πριν από λίγα χρόνια ήταν μονάχα 58. Γιατί υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι φεύγαν σε πρόορη συνταξιοδότηση. Τα πράγματα λοιπόν έχουν βελτιωθεί. Και έχουμε επίση και κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό στη Γαλλία, ότι έχουμε μια δημογραφική ανάπτυξη η οποία είναι θετική. Αν σήμερα λοιπόν έχουμε δυσκολίε για να χρηματοδοτήσουμε το συνταξιοδοτικό μα σύστημα, ξέρουμε ότι σε 10, 15, 20 χρόνια θα είναι μικρότερε οι δυσκολίε λόγω τη ε, δημογραφική αύξηση στη Γαλλία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με άλλε χώρε και οι άλλε χώρε θα πρέπει να έχουν μια ακόμα πιο προσεκτική πολιτική για να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του συνταξιδοτικού συστήματο. Σα ευχαριστώ, κύριε Φεραίρα, τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα σας απευθύνω τις ερωτήσεις στην Πορτογαλική. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντά σας για τις επιτυχίες που έχει δρέψει η Γαλλία πρόσφατα στον οικονομικό στίβο. Μας εξηγήσατε ορισμένες από αυτές τις επιτεύξεις, αλλά η Γαλλία πάντα είχε τη φιλοδοξία να είναι μία από τις ατμομηχανές της Ευρώπης, ένας από τους κύριους παράγοντες της οικοδόμησης της Ευρώπης. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό ποια είναι κατά την άποψή του τα συμπεράσματα που μπορεί να αντλήσει η, η Γαλλία σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα μέσα μια συζήτηση για το ποιο πρέπει να είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και εδώ το ερώτημά μου είναι τι μπορεί να φέρει η Γαλλία με τη δική της εμπειρία για να μπορέσουμε να ξαναθέσουμε την ευρωπαϊκή πορεία σε ένα πιο σταθερό δρόμο. Ένα δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το ρόλο της Ελλάδος. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη αρχίζει να ξαναπαίνει μια δυναμική ανάπτυξη και σταθερότητα, αλλά η Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται και σε επίπεδο Συμβουλίου. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχει εκεί μια θετική αντιμετώπιση ή όχι. Ένα ερώτημα έχει να κάνει με τον φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη που αναφερθήκατε ήδη στο θέμα αυτό και εσείς ο ίδιος. Εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε δημιουργήσει μια ειδική επιτροπή τάξη για τα φορολογικά θέματα και το φορολογικό ανταγωνισμό, σε ποιο βαθμό η, το Συμβούλιο και φυσικά και η Γαλλία στα πλαίσια του Συμβουλίου μπορούν να συμβάλλουν στο να καταλήξουμε σε μια πιο εξισορροπημένη κατάσταση για τη φορολογία στην Ευρώπη και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να περιμένουμε μια πιο εντατική συνεργασία μεταξύ Κομισιών, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά που να είναι σε ένα πιο σοβαρό επίπεδο και αυτό προ όφελο και των πολιτών. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητάμε μεγάλε θυσίε από του πολίτε, ιδίω ορισμένων χωρών, ενώ άλλε χώρε ακολουθούν αυτή την επιθετική φορολογική πολιτική πολιτική που ουσιαστικά αφαιρεί φορολογικούς πόρους από τις χώρες που χρειάζονται αυτούς τους πόρους για την ανάκαμψή τους. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσία σας και για τις απαντήσεις που προσδοκώ. Τρεις ερωτήσεις στο ίδιο κουτί. Θα ξεκινήσω ανάποδα για τα θέματα τα φορολογικά. Είπα ποια είναι η αποφασιστικότητα της Γαλλίας. Η αντίστοιχη υπάρχει και στη Γερμανία και την Ιταλία και σε πολλές ε, μεγάλες χώρες. Ήδη από το 2015 για να είναι εφαρμόσιμο το 2016 θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις έτσι ώστε να τερματιστούν ανώμαλες ζημιογόνες καταστάσεις. Ζημιογόνες σε επίπεδο κοινωνικό. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να σου ζητάνε σαν πολίτη ή σαν επιχείρηση να πληρώσεις φόρους και να έχεις δίπλα σου αυτούς οι οποίοι γλιτώνουν την πληρωμή των φόρων νόμιμα. Λοιπόν, εκεί θα προχωρήσουμε, κάνουμε βήματα, η Επιτροπή θα κάνει προτάσεις, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα ληφθούν αποφάσεις και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ένα συνολικό πακέτο για τα θέματα της αποφυγής φορολογίας. Για την Ελλάδα. Η Γαλλία πήρε μία θέση εξ αρχής και γύρω από τη θέση αυτή περιστρέφονται οι συζητήσεις σήμερα. Αυτό διαπιστώνουμε. Ξέρετε ότι υπήρξε μια ισχυρή αλλαγή στην Ελλάδα ε, σε επίπεδο κυβερνητικό και πρέπει να γίνει σεβαστή. Είναι η αρχή της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τίποτα δεν αλλάζει στις σχέσεις με τους θεσμούς. Είναι θεμητό να ληφθεί υπόψη η εναλλαγή αυτή και να ληφθεί υπόψη η βούληση του ελληνικού λαού. Παράλληλα όμως με αυτό και όχι αντιθετικά με αυτό η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ευρώ. Η κεντρική της τράπεζα είναι η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είναι μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το 1945. Πρέπει λοιπόν να σεβαστεί και τις υποχρεώσεις της. Επί τη βάση αυτών των δύο διαπιστώσεων και αρχών λοιπόν συνεχίζονται οι λύσεις και φυσικά θα βρεθεί λύση γιατί η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας είναι στο ευρώ. Τώρα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Φυσικά και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Οι δυσκολίες που συναντήθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν πολλές και οι ελληνικές αλλά όχι μόνο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στο οικονομικό κομμάτι και το νομισματικό κομμάτι. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε βήματα για να μειωθεί αυτή η έλλειψη ισορροπίας. Μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να χρειαστεί στην παρούσα φάση να αλλάξουμε τις συνθήκες. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία σύγκλησης, εκμεταλλευόμενη τις υπάρχουσες διατάξεις. Οι συζητήσεις θα γίνουν και εδώ, σε εσάς οι, οι σκέψεις τις οποίες οι αποφάσεις σας είναι σημαντικές για μας στον φορολογικό σαν παράδειγμα τομέα ή στον δημοσιονομικό τομέα. Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει και γίνεται ήδη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα γίνει και στο Συμβούλιο για να προχωρήσουμε στα θέματα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Thank ευχαριστώ. Και όντως προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Είναι πολύ αυτή η στάση και η αλλαγή στάση. Σας ευχαριστούμε, Ελίζα, για την ερώτηση αυτή. Ο κύριος Λουκέ έχει το λόγο από την ομάδα του ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ, που ήρθατε εδώ σε εμάς σήμερα. Η γαλλογερμανική φιλία ιστορικά αποτελούσε πάντα την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά θετικά πετύχαμε γιατί ήταν τόσο στενή αυτή η σχέση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Τώρα αυτή η σχέση τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι θολώνει κάπως και ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ε, παραθέτει τον κύριο Σόιμπλε και παραθέτω μια παράδεκτη και αντιπαραγωγική ε, στάση μίσους προς την ε, Γαλλία. Αυτό αντιλαμβάνεται. Αυτά δεν θα τα περίμενε κανείς από δεκαετίες φίλιας. Και ο λόγος ήταν ότι ο κύριος Σόιμπλε είχε δηλώσει ότι το Γαλλικό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να υποχρεωθεί να λαμβάνει τις αποφάσεις που ο κ. Σόιμπλε θεωρεί σωστές. Όντως, η, γαλλική οικονομική πολιτική έλαβε αποφάσεις οι οποίες κινούνται στο περιθώριο των όσων η Ευρώπη έχει συνηθίσει σήμερα. Το τμήμα των ε, γαλλικών επενδύσεων στο ΑΕΠ είναι νομίζω το δεύτερο πιο υψηλό σε όλο τον ΟΣΑ και το, τα κοινωνικές δαπάνες, ε, το ποσοστό κοινωνικών δαπανών της, του ΑΕΠ είναι το πιο υψηλό στον ΩΣΑ στη Γαλλία. Αυτό παράλληλα με ένα έλλειμμα το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να ελεγχθεί από την γαλλική κυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ενδεχομένως ότι υπάρχει μια επιθυμία να εξαναγκαστεί σε κάποια πράγματα η Γαλλία για να υπάρξει μια χρηματοπιστωτική δημοσιονομική εναρμόνιση στην Ευρώπη, αν αυτό επιθυμούμε. Το θέμα είναι όμως αν αυτό μπορεί να συνάδει με κάποιες δημοκρατικές αρχές. Ε, μήπως κάθε λαός θα έπρεπε να μπορεί να λαμβάνει στην Ευρώπη τις αποφάσεις που θεωρεί σωστές ε, για μια κοινωνική εξασφάλιση να έχει την, ε, το δικαίωμα να δεχτεί μια πιο αργή ανάπτυξη. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής δεν πιστεύετε ότι θα ήταν σωστό να τετριθεί αυτή η εθνική κυριαρχία της Γαλλίας και ότι αυτή η επιθυμία με τη γαλλική, και γαλλική κυριαρχία είναι αντίθετη με την περαιτέρω εναρμόνιση στο ευρώ και για την μεγαλύτερη επιρροή στη δημοσιονομική πολιτική των μονομένων κρατών. Δεν είναι αντίθετα αυτά. Ε, <coughs> μα αυτή είναι η Ευρώπη, λέει ο κύριο Σαπέν. Πρέπει σε κάθε μια από τι χώρε μα να κάνουμε αυτό το οποίο είναι καλό για τη χώρα αυτή. Αλλά με το σεβασμό πάντα τη εθνική κυριαρχικότητα. Γιατί η εθνική κυριαρχία είναι και αυτό το τμήμα των συνθήκων. Μιλήσατε για τη φορολογία. Αυτή τη στιγμή είναι πλήρω η φορολογία στα πλαίσια τη εθνική αρμοδιότητα. Αλλά για άλλα θέματα και για θέματα όπω είναι τα θέματα του προπολογισμού και εκεί ο προπολογισμό ψηφίζεται από κάθε εθνικό κοινοβούλιο με συζητήσει, ε, με μια κοινή εποπτεία γιατί βρισκόμαστε στο ίδιο νόμισμα, στο ίδιο οικονομικό σύνολο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τι γίνεται γύρω μα. Αυτό που είναι απαραίτητο όμω στην Ευρώπη είναι για να λειτουργήσει καλά είναι ο σεβασμός τη ε, κυριαρχικότητα κάθε χώρα και των αποφάσεων που λαμβάνονται από κάθε λαό μέσα στα πλαίσια μια αλληλεγγύη. Οι μεταρρυθμίσει που κάνουμε λοιπόν στη Γαλλία δεν είναι κάτι που προέρχεται από τη συζήτηση μεταξύ τη Γαλλία και τη Γερμανία. Φυσικά δεν τα κάνουμε επειδή μα υποχρεώνει κάποιο. Τα κάνουμε γιατί πρώτον είναι καλέ μεταρρυθμίσει αυτέ για τη Γαλλία. Δεύτερον, ξέρουμε γιατί θα είναι καλέ για την Ευρώπη ω σύνολο. Και δεν ιεραρχώ το ότι είναι καλό για τη Γαλλία, τι είναι καλό για την Ευρώπη. Και τα δύο πρέπει να συμβαδίζουν. Το ότι η Γαλλία θα πρέπει να μειώσει τα ελλείμματά της και να σεβαστεί τι υποχρεώσει τη είναι καταρχήν καλό για την ίδια τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν μπορεί να συσσωρεύει χρέη και ελλείμματα χωρί προβλήματα. Οι αγορέ μα την, δίνουν την εμπιστοσύνη του, μα δανείζουν χρήματα με το ίδιο σχεδόν επιτόκιο όπω στη Γερμανία και σε άλλε χώρε, αλλά θα πρέπει να αξίζει κανεί την εμπιστοσύνη των αγορών. Αλλά οι πράξει μα επίση ε, έρχονται και από την αλληλεγγύη προ τι άλλε χώρε τη Ευρώπη και τη Ευρωζώνη. Μια χώρα όπω η Γαλλία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο προέρχεται από την ιστορία, αλλά και η πραγματικότητα τη Ευρώπη τη δίνει αυτό το ρόλο και αυτή την ευθύνη, μια ευθύνη όχι μόνο απέναντι στον εαυτό τη, αλλά απέναντι και σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θέλω η Γαλλία να αναλάβει τι ευθύνε τη, έναντι του δικού τη λαού, αυτό είναι ευθύνη τη κυβέρνηση και του Κοινοβουλίου για τον γαλλικό λαό, αλλά θέλω η Γαλλία να αναλάβει και τις ευθύνε της και να είναι στο ύψο των ευθυνών τη και απέναντι σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Και αυτό ξεπερνάει απλώ το γαλλο-γερμανικό διάλογο. Μερικές φορέ βλέπει κανεί στο γερμανικό τύπο τις δηλώσεις του α ή β αξιωματούχου μέσα στο α ή β κόμμα. Αυτά μπορεί να είναι αρνητικά ή δυσάρεστα για τη Γαλλία. Αυτό είναι το τμήμα τη συζήτηση. Αλλά και στη Γαλλία πολλέ φορέ γίνεται κάτι αντίστοιχο για τη Γερμανία. Μπορώ να σα πω όμω το εξή ποτέ δεν μπορεί να επιληθεί τίποτα στην Ευρώπη αν υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και αν θέλετε να το πω και θετικά, τίποτα το ουσιαστικό δεν μπορεί να γίνει στην Ευρώπη αν δεν υπάρξει σύγκληση απόψε μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και δεύτερον, αυτό είναι μια δεύτερη σημαντική προϋπόθεση, αν αυτή η σύγκληση απόψεων μπορεί να έχει και την σύμπραξη των άλλων. Αν δεν είναι μια συμφωνία η οποία μπορεί να την εγκολποθεί και το υπόλοιπο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η απόψή μου για το γαλλογερμανικό διάλογο και εγώ τα καταφέρνω πολύ καλά. Έχω πολύ καλή ε, συνεννόηση με τον κύριο Σόιμπλε, ακόμα και αν πει κάποια λόγια τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν ως ε, δυσάρεστα. Πάντα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μα. όταν είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Η κυρία Κόρα από την Άλτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα το ότι ήρθατε εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα καταρχάς να θέσω το θέμα του μανιφέστο του Σοσιαλιστικού Κόμματος που παρουσίασε κύριε Δέλη, το οποίο υποστηρίξατε και εσείς. Το μανιφέστο λοιπόν αυτό καλεί μεταξύ άλλων και για μια χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και η ΕΚΤ να καταστεί ε, τελικό καταφύγιο πίστοσης για τους ε, για τις χώρες. Καταγνωρίζετε την σημασία των κοινών δημοσιονομικών κανόνων για να υπάρχει κοινή ε, πολιτική δημοσιονομική στην Ευρώπη και συμφωνείτε με το μανιφέστο που ζητάει την ε, γενικότερη χαλάρωση και πιστεύετε ότι το, το κείμενο του μανιφέστο θα χρησιμεύσει προκειμένου να διασφαλίσει και να εξασφαλίσει και να πείσει τις άλλες χώρες ότι η Γαλλία θα μείνει στα συμφωνημένα όρια για την οικονομία της και για την ε, συνεργασία την επικοδομητική με τους Ευρωπαίους εταίρους και κατά δεύτερον να σας ρωτήσω για το οικονομικό πακέτο, το νομοθετικό πακέτο οικονομικών μεταρρυθμίσεων Λουά Μακρόν, όπως αυτό α, ονομάζεται ο κύριος Μακρόν και παραθέτω είπε ότι κάποιοι σκληροί στο Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν θα πρέπει να μπορέσουν να αλλάξουν την πορεία μαζί τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Συμφωνείτε με τον συνάδελφό σας ότι χρειάζεται μια σκληρή στάση, ιδιαίτερα στη φάση εφαρμογής του νόμου και σε ό,τι αφορά το ελεύθερο ωράριο. Συμφωνείτε ότι το υψηλό φορολογικό, η υψηλή φορολογική επιβάρυνση, η Δαπάνε του κράτου, όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μεγάλη επιβάρυνση. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα και ευχαριστώ που παρακολουθείτε τόσο προσεκτικά τις εσωτερικές συζητήσεις του κόμματο. μου. Και εγώ θα παρακολουθήσω με την αντίστοιχη προσοχή το τι κάνετε εσείς στο δικό σας κόμμα και θα κοιτάξω όλα τα κείμενα τα οποία θα προτείνουν τα μέλη σας. Ε, θα είναι μια καινοτομία για μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ και για το χαμόγελό σας. Να πω ότι οι ερωτήσεις σας ήταν απολύτως θεμητές. Η Γαλλία οικοδόμησε μαζί με άλλους συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες και μαζί με άλλους και μαζί με άλλες χώρες ε, ε, έβαλε μέσα και συγκεκριμένες μορφές ευελιξίας. Η Γαλλία θέλει τον σεβασμό των κανόνων, με μια κάποια ευελιξία η οποία ήδη εμπεριέχεται στους κανόνες. Και σε αυτό το πλαίσιο ελήφθησαν και οι αποφάσεις και της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τη Γαλλία, ιδιαίτερα η τελευταία σύσταση του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως γνωρίζετε και το παρατηρήσατε η σύσταση αυτή είναι απολύτως συγκλίνουσα για πρώτη φορά με τις αποφάσεις τις οποίες πήρε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και με τις προβλέψεις τις οικονομικές που είχε πάρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη Τρίτη. Λοιπόν, για αυτή τη σύγκληση ε, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να μην υπογραμμίζουμε κάποια επιμέρους αποκλίνοντα στοιχεία. Τώρα για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, επαναλαμβάνω, απαραίτητες και για τη Γαλλία, Μιλήσατε για το άνοιγμα των καταστημάτων ε, την Κυριακή, στις τουριστικές περιοχές. Αυτό είναι προφανές. Έρχονται τουρίστες ε, τις Κυριακές, τη Δευτέρα φεύγουν. Αν ε, δεν αγοράσουν την Κυριακή θα πάνε σε άλλη χώρα να αγοράσουν τη Δευτέρα. Λοιπόν, προφανώς θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες διεθνείς οικονομικές ζώνες στη Γαλλία που θα είναι ανοιχτές την Κυριακή. Αυτό προκαλεί συζητήσεις. Ε, αυτό προκαλεί συζητήσεις και στην κυβερνητική πλειοψηφία. Εσείς αναφερθήκατε ε, στη χρήση ενό όπλου που δίνει το Σύνταγμα στη γαλλική κυβέρνηση, το νόμο 49 κάθετος 3. Τον χρησιμοποιήσαμε τον νόμο αυτό για να υιοθετήσουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε, πάνω σε αυτά υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία πάντα οι αποφάσεις διαμορφώνονται από την πλειοψηφία κάθε φορά. Στο συγκεκριμένο θέμα υπήρξε μία κάποια δυσκολία και μία κάποια καθυστέρηση. Δείξαμε ότι ήμασταν αποφασισμένοι πάντως γιατί θέλαμε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση, εμείναμε στη μεταρρύθμιση και μέχρι την τελευταία στιγμή θα αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδημούλης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Σαπέν, σας καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται θάρρος, όπως είπε ένας Γερμανός συνάδελφος, για να είσαστε εδώ. Η ομιλία σας ήταν ένα ύμνος στην ανάγκη να αναζητούμε συμβιβασμούς, γιατί έτσι μόνο μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη, στην ανάγκη να μελετούμε και τις κοινωνικές συνέπειες των μεταρρυθμίσεων, και να αναζητούμε και την σταδιακότητα που θα επιτρέπει την εξασφάλιση της αναγκαίας συνένεσης. Είπατε ότι η Γαλλία εξασφαλίζοντας αυτήν την ελαστικότητα και ευελιξία στην ερμηνεία του Συμφώνου της Σταθερότητας ήδη έχει κάποια θετικά σημάδια για την οικονομία. Είμαι βέβαιος ότι αυτή την ελαστικότητα δεν την θέλετε εσείς προσωπικά μόνο για τις μεγάλες χώρες αλλά για όλες τις χώρες σημείωσα με ικανοποίηση και αυτό που είπατε ότι είναι ανάγκη ε, στο Συμβούλιο, στο Eurogroup να πάρετε υπόψη, να ληφθεί υπόψη η ισχυρή βούληση των Ελληνίδων και των Ελλήνων για αλλαγή και αυτό να συνδυαστεί με ένα συμβιβασμό με την ανάγκη σεβασμού των κανόνων. Συμφωνώ μαζί σας η κυβέρνηση, η νέα η ελληνική θέλει αυτό το συμβιβασμό, εργάζεται για αυτό το συμβιβασμό. χθες υπήρξε μια κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού Τσίπρα με τον πρόεδρο της Κομισιόν που ανοίγει δρόμο για αυτό το συμβιβασμό γεφυρώνοντας διαφωνίες σε σημεία αγκάθια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αποφάσεις του στην προηγούμενη θητεία έχει μιλήσει με πολύ αυστηρή κριτική για τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες που προκάλεσε το μνημόνιο και η τρόικα στην ελλάδα εγκρίνοντας εκθέσεις με μεγάλη πλειοψηφία η ερώτησή μου είναι μία σαφής και συγκεκριμένη τι περιμένετε να γίνει στο Eurogroup της 11ης Μαΐου που να υποβοηθά και να επιταχύνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί τις δύο, τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να απαντηθεί το οξύ πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δημόσια οικονομικά μέχρι ότου οικοδομηθεί η συμφωνία και τρίτον τι θα κάνετε εσείς προσωπικά συμβάλλοντας σε αυτό το συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σταματήσω εκεί θα ξεκινήσω μάλλον από εκεί που ε, ξεκινήσατε και εσείς ο ίδιος κύριε Βουλευτά. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Είναι ήδη για όλους. Σε ό,τι αφορά το σεβασμό των κανόνων δεν υπάρχουν μεγάλες ούτε μικρές χώρες. Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν μεγαλύτερο οικονομικό ειδικό βάρος στη ζωή του ευρώ. Αυτό είναι προφανές. Αυτό το οποίο γίνεται σε μια χώρα η οποία έχει ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 30% ή 20% είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πάντα μα ενδιαφέρει και αυτό που γίνεται σε σχέση με την εξέλιξη του ΑΕΠ στην, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου υπήρξε τεράστια απώλεια του ΑΕΠ, κάτι το οποίο είχε πολύ οδυνηρέ συνέπειε για τον πληθυσμό τη Ελλάδος και δημιούργησε μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη και οδυνηρή και φυσικά και πολιτικά ιδιαίτερα ευαίσθητη. Οι όμω. με την ευελιξία που περιλαμβάνουν είναι ήδη για όλου. Και η Ελλάδα είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που αντιμετωπίζεται με κάποιο τρόπο, για να το πω έτσι ουδέτερα από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, υπάρχουν συνοδευτικές προσπάθειες από τις χώρες του ζώνης του ευρώ που τη βοήθησαν να περάσει τα τελευταία δύσκολα χρόνια και να αντιμετωπίσει μια σειρά από προθεσμίες και συνεχίζει αυτή η διαδικασία και θέτεται το ερώτημα για τι επόμενε εβδομάδε. Ίσως αυτό θα συνεχίσει και επέκεινα τις επόμενε εβδομάδες. Η Ελλάδα λοιπόν ίσω θα χρειαστεί να έχει την υποστήριξη τη ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όμω υπόκειται σε ορισμένου κανόνε. Και το είπατε και εσεί ο ίδιο ότι αυτοί οι κανόνε θα πρέπει να τύχουν σεβασμού και από την ελληνική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι είναι και η θέληση τη ελληνική κυβέρνηση να το πράξει και Είμαι πεπισμένο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Θα σα δώσω τη δική μου άποψη τώρα για τα θέματα αυτά και θα απαντήσω στο ερώτημα που θέσατε για την 11η Μαου, δηλαδή για τι συνεδρίε του Eurogroup την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει η ευελιξία. Προφανώ η ελληνική κυβέρνηση, το μεγαλύτερο μέρο τη ελληνική κυβέρνηση, έχει τη θέληση να αλλάξει κάποια στοιχεία του προγράμματο αυτού. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν αυτά τα στοιχεία που θα αλλάξουν με άλλα στοιχεία ώστε η συνολική ισορροπία σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο προπολογισμού να γίνει σε Είναι η συνολική ισορροπία του προγράμματος και του προπολογισμού που θα πρέπει να διατηρηθεί ώστε η αλληλεγγύη και η υποστήριξη από την υπόλοιπη Ευρωζώνη και Ευρώπη να διατηρηθεί. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή την ισορροπία να διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει που δεν μπορούμε να αλλάξουμε με μονομένα στοιχεία σε συνάρτηση με τη θέληση τη ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η τροποποίηση θα πρέπει να γίνει με αντιστάθμιση των στοιχείων που αλλάζουν με άλλα αντίστοιχα στοιχεία. Παραδείγματο σε ό,τι αφορά την ε, ε, φορολογία ή την συμμετοχή στον προπολογισμό τη ε-, Ελλάδο από διάφορε πτυχέ. Εδώ τώρα δεν για την 11η Μαΐου. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι το οριστικό ορόσημο. Εγώ πιστεύω όμως ότι η 11η Μαΐου θα πρέπει να είναι και το ελπίζω και το πιστεύω μια θετική ημερομηνία που θα δείξει τα πράγματα προχωρούν θετικά και επομένως ο δρόμος προς μια συμφωνία θα είναι ο δρόμος που θα έχουμε να διατρέξουμε και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνο ενό ατυχήματο μέσα σε εισαγωγικά ή μια αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Θέλουμε όλοι λοιπόν η 11η Μαΐου να είναι μια θετική χρονική στιγμή, να υπάρχει το θετικό κλίμα, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή τη θετική πορείας, ώστε όλοι και οι μεν και οι δε να μπορέσουν να βρουν μια καλή συμβαστική λύση, να υπάρξει συμφωνία για το πρόγραμμα αυτό, αλλά να υπάρξουν και θετικές διέξοδοι για το μέλλον μετά από αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Δέκα ομιλητές έχω ακόμα. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα 48 λεπτά που μας μένουν, ώστε να μπορέσουν όλοι να λάβουν, θα πρέπει οι ερωτήσεις να περιοριστούν ε, σε λιγότερο από 5 λεπτά και δίνω καταρχήν το λόγο, μαζί με την απάντηση, σε λιγότερο από 5 λεπτά, δίνω καταρχήν το λόγο στην Εύα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό που είναι μαζί μας σήμερα και που μοιράζεται μαζί μας τις ανησυχίες του. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω κάπως καλύτερα τη θέση της Γαλλίας στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Συνειδητοποιούμε την σημασία της θέσης της Γαλλίας και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμένουμε τόσο πολύ στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Ενώ η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα προτείνει την καταπολέμηση της διαφθοράς, την καταπολέμηση των απατών. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτός ο αγώνας θα είναι πιο χρήσιμος για την επανεξισορρόπηση των ελληνικών δημοσιονομικών από ότι η μεταρρύθμιση βράχει πρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα της αγοράς εργασίας. Θα εμείνετε σε αυτή τη μεταρρύθμιση, ενώ στα σύνορα της Ευρώπης έχουν ξεσπάσει μεγάλες πυρκαγιές Νομίζω ότι η παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι μια εγγύηση σταθερότητας για την ίδια την Ευρώπη και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι μια χώρα η οποία διοικείται με άσχημο τρόπο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ε, είναι μια από τις χώρες με φαινόμενα ισχυρότατα διαφθοράς και αυτή η πλήρης απελευθέρωση θα οδηγήσει φοβάμαι σε ε, μεγαλύτερη εξαέρωση των φορολογικών εσόδων. Μια δεύτερη ερώτηση τώρα αφορά την καταπολέμηση ε, της φοροαποφυγής ε, και, της, και αντίστοιχα φαινόμενα και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα μεγάλων επιχειρήσεων και μάλιστα έχουμε και επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα ε, στον τομέα τον εξορυκτικό που δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα ή πληρώνουν κάτι συμβολικά ποσά ενώ ε, οι χώρες αυτές έχουν την έδρα τους στη φορολογική στην Ολλανδία. Πρόκειται για κάποια σχήματα, για κάποια προγράμματα πάρα πολύ ε, τεχνητά και αρνητικά. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε πληροφορίες για τις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις, το τι συμβαίνει όπως το κάνετε για τις τράπεζες. Έχουμε κάνει τέτοια τεστ αντοχής ε, για τις τράπεζες, είδαμε το τι συμβαίνει, πρέπει να το δούμε και για τις μεγάλες ε, διεθνείς επιχειρήσεις. Τώρα υπάρχει και το άλοθη της αποφυγής της χρήσης της μεθόδου της διπλής επιβολής. Αυτό επιτρέπει σε πολιεθνικές να μην πληρώνουν πουθενά ε, φόρο. Ευχαριστώ κύριε Σολή. Μετά από τρία λεπτά έχουμε μόνο δύο λεπτά για απάντηση. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να το πιο σύντομο στην απάντηση. Είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό για την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχουν αναφερθεί και όλε οι προτάσει οι οποίε γίνονται αυτή τη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συλλογή των φορολογικών εσόδων. Προφανώ πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά τα οποία θα επιτρέψουν να ενισχύσουμε ή να δημιουργήσουμε καλύτερα φορολογικέ διοικήσει που θα είναι αποτελεσματικέ και έντιμε είναι πάρα πολύ σημαντικό ήταν ένα από τα στοιχεία των προηγουμένων συμφωνιών και ήταν ένα στοιχείο το οποίο δεν είχε εφαρμοστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να αποθαρρύνουμε την ελληνική κυβέρνηση από το να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και η Γαλλία είναι έτοιμη και με μια συνεργασία σε επίπεδο διοικητικό να βοηθήσει την Ελλάδα να δημιουργήσει συστήματα τα οποία είναι αποτελεσματικά στο φορολογικό χώρο. Για την αγορά εργασίας το βασικό θέμα δεν είναι το θέμα της ε, αγοράς εργασίας όσο η πρόταση για τον ελάχιστο μισθό σε ε, επίπεδο διαπραγματεύσεων. Καταλαβαίνουμε την πρόθεση της Ελλάδος να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, αλλά ο ρυθμός αύξησης αυτού του κατώτατου μισθού προφανώς θα έχει επιπτώσει στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αυτό το θέμα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ίσως είναι πιο δύσκολα για τον αγώνα κατά της φόρο αποφυγής δεν Δυσκολεύομαι να σας πω ότι αυτό είναι το κύριο θέμα της σημερινής συζήτησης. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία έχουν πάρει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και μέσα στο 2015 έχουμε αποτελέσματα που θα μας επιτρέψουν από του χρόνου να τεθούν όλα αυτά τα μέτρα ε, σε εφαρμογή. Ναι, θα πρέπει το θέμα της διπλής φορολόγησης να αντιμετωπιστεί γιατί δεν θα, επιτρέπει, δεν θα πρέπει να επιτρέπει την μη φορολόγηση καθόλου και από τις δύο πλευρές. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και είναι απαραίτητο μέχρι το τέλος του χρόνου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα για το θέμα αυτό. Και τέλος. Για την συνεργασία των χωρών θα πρέπει να γίνει καταρχήν μεταξύ διοικητικών αρχών και θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει και στη συνέχεια περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών. Πέντε λεπτά λοιπόν ε, για ερώτηση και απάντηση ο κ. Δεβάλη. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό που είναι παρόν και δίδει απαντήσεις. Θα είμαι συνοπτικότατος. Στα πλαίσια του Working Group για την αναθεώρηση της διακυβέρνησης, οι θέσεις οι γίνονται δεκτές από πολλές χώρες, ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους μηχανισμούς αλληλεγγύης και την νομιμοποίηση τη δημοκρατική της διαδικασίας. Τα υπόλοιπα όμως είναι λίγο θολά. Μιλάτε για απλοποίηση του εξαμήνου ας πούμε. Τι θα πει αυτό. Ε, Πάντως υπάρχουν φήμες ότι το Βερολίνο και το Παρίσι θα προτείνουν ένα οδικό χάρτη πριν από τα μέσα του καλοκαιριού για την οικονομική διακυβέρνηση. Μπορείτε να συνδυάσετε τις θέσεις σας με τους Γερμανούς. Εσείς στη Γαλλία ζητάτε να υπάρξει μια περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα συνδυαστείτε με τις αντίστοιχες γερμανικές θέσεις. Και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ε, στον γαλλικό προϋπολογισμό μιας πιθανής εξόδου από την Ευρωζώνη της Ελλάδας. Για την τελευταία σας ερώτηση, ε, δεν κάνω κανένα τέτοιο υπολογισμό, γιατί η θέση της Ελλάδας είναι μέσα στο ευρώ. Και η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ. Πρώτον γιατί αυτό το επιθυμεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός γιατί αυτή είναι η εκπεφρασμένη επιθυμία της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Ελλάδα και γιατί η δυναμική της Ευρώπης δεν είναι να αυτομοιούται αλλά να διευρύνεται και θα ήταν μια πολιτική αποτυχία και δεν μιλάω για τα οικονομικά θα ήταν μια πολιτική αποτυχία αν ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο από τον δρόμο της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ. Τώρα στα υπόλοιπα. Η κατάσταση σήμερα είναι διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν. Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι μηχανισμοί βοήθειας προς τα πιστοτικά ιδρύματα και προς τα κράτη-μέλη και δεν θα δημιουργηθούν τεράστιες δυσκολίες και γι' αυτό συγκεντρώνουμε την προσοχή μας, επαναλαμβάνω, στην επιτυχία του παρόντος διαλόγου να επιτευχθεί ο συμβιβασμός και η απόφαση για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Τώρα για την μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης. Σας έδωσα κάποια πρώτα στοιχεία. Έχουμε προχωρήσει στον τομέα αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη αντίληψη που να φτάνει μέχρι και την αλλαγή των συνθήκων. Υπάρχει επίσης όπως είπατε μια πρωτοβουλία γαλλογερμανική. Είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε. Αλλά όπως είπα θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική, ολιστική αντίληψη της δημοσιονομικής κατάστασης και στον κοινωνικό τομέα και στον οικονομικό τομέα στην Ευρώπη. Και μετά, ανά χώρα, θα προχωρήσουμε στις συστάσεις που είναι απαραίτητες για τις χώρες μας. Thank you. Now, Mr. Bernard Ο κύριος Μονό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Η Γαλλία είπε ότι θα έχει μηδενικό έλλειμμα το 2017. Είναι πολύ μακριά αυτός ο στόχος τη στιγμή που είμαστε στο 3,8 αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρείτε 4 δισεκατομμύρια ευρώ στον ε, εξοικονομήσεις στον ε, προϋπολογισμό σας, όπως ζήτησε ο κύριος Μοσκοβισή, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε ιστορικά χαμηλά επιτόκια στις αγορές αν φτάσουν τα επιτόκια ε, στο 1% το βάρος της Γαλλίας θα αυξηθεί κατά 10 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα συνολικό βάρος 220 δισεκατομμύρια ε, ευρώ και προσπαθείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή ε, περισσότερα χρήματα με το να αυξάνετε το κοινωνικό βάρος και αυξάνοντας τις, το βάρος του εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί το βάρος των εργαζομένων και αυτό χωρίς να λάβουμε υπόψη τις πρόσθετες χρηματοδοτικές εγγυήσεις που οδήγησαν σε μεγάλη λιτότητα. Οι φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες λύσεις λοιπόν δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, θα καταλυστεύσουν την, την οικονομία της Γαλλίας και δεν ανταποκρίνονται σε κανένα πατριωτικό αίσθημα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύσετε το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσετε πολύ καλά τι σημαίνει το τι σημαίνει να δημιουργούνται χιονοστιβάδες. Αν σύμφωνα με την ε, έκθεση της, ε, της Τάπεζας Γαλλίας ξεπεραστεί το όριο αυτό, τι θα γίνει. Εσείς θέλετε να έχετε ένα εξισορροπημένο προπολογισμό, αλλά με ποιο τρόπο θα αρχίσετε να ξεπληρώνετε τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ του γαλλικού χρέου. Και επίση, προβλέπετε να υπάρξει έλεγχο φορολογικό των μεγάλων γαλλικών εταιριών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του LuxLeaks. Σα ευχαριστώ για την απάντησή ε, είναι πάρα πολύ επακριβή η ερώτησή σα, οπότε εγώ θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ εξίσου ακριβή. Δεν κατάλαβα τώρα αν εσείς υποστηρίζετε τη μείωση των δημοσίων δαπανών και των ελλημάτων ή αν τα κατακρίνετε αυτά. Η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει μια προοπτική να μειώσει κατά 50 δισεκατομμύρια τις δημόσιες δαπάνες μέχρι το 2017, για τα τρία αυτά χρόνια, το 2015-2017. Με αυτή τη μείωση των δημοσίων δαπανών θα μπορέσουμε μεν να χρηματοδοτήσουμε βασικές προτεραιότητες όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η εξωτερική και η εσωτερική ασφάλεια, αλλά με τις εξοικονομήσεις των 50 δισεκατομμυρίων αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και μείωση των φορο, της φορολόγησης όχι μόνο των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων και θα μπορέσουμε επίσης να μειώσουμε και το έλλειμμα του προϋπολογισμού μας για να μειώσουμε και το χρέο μα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Δεν είναι η Κομισιόλη λοιπόν, που σα ε, υποχρεώνει να κάνετε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια εξοικονομήσεων. Είναι απαραίτητε εξοικονομήσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό που δεσπίσαμε ω κυρίαρχο κράτο και το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε. 21 <clears throat> δισεκατομμύρια εξοικονομήσεων απαραίτητα εφέτο. Θα επιτύχουμε λοιπόν αυτό το στόχο χάρη στα 4 αυτά πρόσθετα δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν απαραίτητα όλα αυτά για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τι υποχρεώσει μα όχι μόνο έναντι τη Ευρώπη αλλά κυρίω έναντι του γαλλικού λαού και του γαλλικού κοινοβουλίου. Αυτή ακριβώ είναι η στρατηγική που ακολουθείται από τη γαλλική κυβέρνηση. Δρούμε υπέρ τη Γαλλία μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο γιατί πιστεύουμε στη σημασία του ευρωπαϊκού πλαίσιου. Κάποια μέρα θα πρέπει να κάνετε και εσείς κάποιο υπολογισμό του τι θα στήχιζε στη Γαλλία να βγει από το ευρώ και θα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν νόημα τα επιχειρήματά σας δεν απαντάτε για το αν θα κάνετε φορολογικό έλεγχο στις μεγάλες γαλλικές εταιρείες που εμπλέκονται στο LuxLeaks. Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Ναι, να συμπληρώσω. Απήντησα και σε άλλους ομιλητές. Θέλουμε να σταματήσει αυτός ο μηχανισμός ε, που αποφυγής της φορολόγησης θέλουμε λοιπόν να υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές των χωρών μας να ξέρουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση σε φορολογικό επίπεδο των εταιριών μας όχι μόνο στο εδαφός τους αλλά και έξω από το εδαφός τους οπότε οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευνοηθεί από συμφωνίες για να μην πληρώνουν φόρους θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερο φόρο στις Γαλλίες. Αυτό λέτε για το μέλλον, αλλά τι θα γίνει για το παρελθόν, αυτά τα χρήματα που έχουν ήδη χαθεί. Ο Ernst, η Ernst Lange έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο ερωτήσει για δύο λεπτά και έτσι τρία λεπτά θα έχετε για να απαντήσετε. Για την γενικότερη συζήτηση που θα θέλετε να γίνει για την Ευρωζώνη στο σύνολό τη. Το καλωσορίζουμε αυτό επί τη αρχή. Θα μπορούσατε να είστε πιο σαφεί όμω, Είπατε ότι θέλετε μια πιο συνολική συζήτηση και μετά να εφαρμοστούν τα μεμονωμένα στοιχεία στα κράτη-μέλη. Αυτό τι σημαίνει. Όσο μια χώρα όπως η Γερμανία έχει ισορροπημένο ισοζύγιο υπολογισμού, προπολογισμού, οι άλλοι μπορούν να πάνε πάνω από το 4%. Πώς φαντάζεστε ότι θα γίνει αυτή η συνολική συζήτηση και πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μόνα μέλη ή μήπως οι κανόνες ισχύουν για όλους με τον ίδιο τρόπο και μετά από τη συζήτηση αυτή. Δηλαδή το 3% ισχύει για όλους με την ίδια ταχύτητα και με τον ίδιο ένταση. Κατά δεύτερον, αν θέλετε να γίνει μια συζήτηση για τη θέση της Ευρωζώνης στο σύνολό τη. δεν μπορεί αυτό να ειδωθεί μεμονωμένα ή να υποκριθούμε ότι η Ευρωζώνη είναι νήσος ε, απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και τη θέση της Ευρωζώνης στην παγκόσμια οικονομία. Και τότε το μόνο που μπορούμε να εξαγάγουμε στο συμπέρασμα είναι ότι χάνουμε ανταγωνιστικότητα. Είμαστε κάτω από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχουμε 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, 50% της ε, παγκόσμιας ε, ευημερίας σε ό,τι αφορά τις δαπάνες κοινωνικής ε, φύσεως. Δηλαδή, με ένα μικρό πληθυσμό που γυράσκει κιόλας, έχουμε μεγάλο τμήμα της οικονομικής ισχύω. Αν θέλουμε να έχουμε μια ευκαιρία να το κρατήσουμε αυτό θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε καινοτομικοί. Γιατί δάλλως να κάνουμε την, την εργασία στην Ευρώπη όσο φτηνή είναι και στην Κίνα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και πιο ανταγωνιστικοί. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η ατζέντα και αυτή θα εκπληρωθεί και στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρωζώνη. Η ερώτηση είναι σύντομη, αλλά παρόλα αυτά ανοίγει πάρα πολλά θέματα. Ξεκινάω από το τέλος πάλι. Θα πρέπει να δείξουμε ευφυΐα, θα πρέπει να δείξουμε καινοτομία, θα πρέπει να δείξουμε ανταγωνιστικότητα. Διακυβεύεται το μέλλον της Υπήρου μας. Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το θέμα είναι πρώτα να σκεφτούμε συνολικά τη ζώνη ευρώ και μετά τις επιμέρους χώρες. Έτσι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν πηγαίνω στην ομάδα των 20, στο G20 ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το βασικό πρόβλημα του κόσμου για πολλούς μήνες ήταν το τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Γιατί είναι τόσο χαμηλή η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, γιατί αυτό έχει επιπτώσεις και στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί υπάρχει τόσο χαμηλός πληθωρισμός στη ζώνη ευρώ, κάτι το οποίο προκαλεί συνέπειες και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν βλέπουν μία χώρα μεμονωμένα. Βλέπουν τη ζώνη ευρώ, βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό πρέπει να σταθούμε κι εμείς. Μέσω των αλλαγών, μέσω της καινοτομίας θα διατηρήσουμε τη θέση της Ευρώπης και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε άλλους τομείς, στον πολιτικό τομέα, τον πολιτιστικό τομέα, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία μιας υπήρου όπως η δική μας. Λέτε πώς θα περάσουμε από τη σφαιρική αντίληψη στις μεμονωμένες περιπτώσεις των χωρών. Αυτό κάνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή κάνει μια ανάλυση της κατάστασης στη ζώνη ευρώ, στο δημοσιονομικό. Και μετά από αυτό θα κάνει προτάσεις αναχώρα και σε χώρες όπως η Γερμανία αυτό. Θα, κάνει, δημιουργήσει συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει πράγματα και στην Γαλλία, λέει πράγματα και στην Γερμανία. Ε, πράγματι υπάρχουν χώρες γιατί έχουν κάνει πράγματα στο παρελθόν, διευκολύνουν τις ξένες επενδύσεις. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα παραδείγματα και να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε όλες τις χώρες για να υπάρξουν αντίστοιχες καταστάσεις σε όλες τις χώρες. Έτσι μόνο η Ευρωζώνη θα σταθεί στο ύψος των ευθυνών της σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί ο κόσμος μας κοιτά, μας βάζει ερωτήσεις, ο κόσμος μας θέλει, θέλει μια Ευρωπαϊκή Ήπειρο η οποία να είναι επιτυχής. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ήπειρος δεν πάει πολύ καλά, ο υπόλοιπος κόσμος ανησυχεί. Κοιτάξτε σε 10 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν άκουσα το πώς η Γαλλία και η Ευρώπη θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα. Πώς πρέπει να μας δώσετε μια απάντηση σε μια άλλη φάση. Στην επόμενη απάντησή σας. Είδατε ότι στις προβλέψεις της Επιτροπής για, την, για τον επόμενο χρόνο ε, ένας από τους λόγους που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη είναι και οι αλλαγές στον τομέα της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Υπάρχουν ε, καλοί λόγοι στην δύσκολη σημερινή κατάσταση για να βρούμε μια ρεαλιστική λύση με την Ελλάδα. Και υπάρχουν και καλοί λόγοι στην τρέχουσα κατάσταση να είμαστε δημοσιονομικά αντικειμενικοί σε ό,τι αφορά το όριο δενικών επιτοκίων, σε ό,τι αφορά μια μεταρρυθμιστική ατζέντα που θα πρέπει να υπάρξει επίσης και να είναι και αλλά παράλληλα η ευέλικτη αντιμετώπιση των κανόνων υποσκάπτει τους κανόνες και καταδεικνύει και τα, συν, τους. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα για το κατά πόσον ε, η στρατηγική που απαντήσατε προηγουμένως μιας ε, βαθμιαίας εξέλιξη των κανόνων θα επαρκέσει προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα και να υποστηριχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του συνολικού συστήματος. Μήπως καλύτερος τρόπος δεν θα ήταν να ξεκινήσουμε τώρα και να εμβαθύνουμε την Ευρωζώνη με μια συνταγματική, μια αλλαγή τροποποίηση της ε, συνθήκης, ενισχύοντας ε, την ε, δημοκρατία. Τι πιστεύετε ότι... Τι ισχύει για μια τέτοια στρατηγική. Σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα και <laughs> ξέρω ότι γνωρίζετε πολύ καλά τη Γαλλία, έχετε θέσει το θέμα αυτό και στα γαλλικά στο παρελθόν. Εγώ δεν πιστεύω. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέσει κανεί ένα τέτοιο ερώτημα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν θεωρώ ότι η ευκαμψία μέσα στην εφαρμογή των κανόνων και για μένα η ευκαμψία είναι κομμάτι των κανόνων. Δεν νομίζω ότι η ευελιξία θέτει ένα αμφιβόλο την αξιοπιστία των κανόνων. Κάθε άλλο. Το αντίθετο. Από πέρσι επειδή ακριβώς μπορέσαμε να είμαστε απαιτητικοί για τη μείωση των ελλημάτων, αλλά πιο πραγματιστικοί και πιο ευέλικτοι στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, γι' αυτό η Ευρωζώνη πηγαίνει πολύ καλύτερα. Και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήρε σημαντικές αποφάσεις. Τελικά έχουμε καταλήξει να είμαστε πιο αξιόπιστοι σε σχέση με τον εξωκόσμο. Πέρσι τον Οκτώβριο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν η Έλα κάνει την ανάλυση των κινδύνων σε όλο τον κόσμο, τότε θεωρούσε ως πρώτο κίνδυνο την Ευρωζώνη. Πριν από λίγες μέρες συναντηθήκαμε πάλι στη Ουάσιγκτον. Ο κίνδυνος της Ευρωζώνης είχε εξανεμιστεί. Επομένως η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης είχε ενισχυθεί γιατί υπήρξε ευφυής εφαρμογή των κανόνων που είναι οι κανονισμός. Θα έπρεπε να προχωρήσουμε περισσότερο για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ναι, θα έλεγα. Θα πρέπει να έχουμε μια δυναμική εμβάθυνση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι την τροποποίηση των συνδικών. Λένε ορισμένοι, το καταλαβαίνω ότι το λένε αυτό. Αυτή τη στιγμή όμω θα ήταν κάπω δύσκολο. Θα θέταμε τον εαυτό μα σε πολύ μεγάλε δυσκολίε και θα μα εμπόδιζε στο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τι απαραίτητε ενέργειε. Πρέπει να τα δούμε λοιπόν σε δύο φάσει. Σε μια πρώτη φάση πρέπει να είμαστε πραγματιστέ, να λειτουργήσουμε με τι τωρινέ συνθήκε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε καλύτερη σύγκληση μέσα στα πλαίσια των συνθήκων που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, θα δούμε στη συνέχεια αν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Αλλά μια συμφωνία για την αλλαγή των συνθήκων πρέπει να έχει και δημοκρατική υποστήριξη. Έχετε απόλυτο δίκιο για το θέμα αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτή από τους λαούς μας μια τέτοια αλλαγή παρά μόνο αν η Ευρώπη πάει καλύτερα σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο απασχόληση, σε επίπεδο φορολογικής δικαιοσύνης. Η πρώτη μας λοιπόν ευθύνη είναι να δώσουμε την εμπιστοσύνη στους λαούς μας ότι η Ευρώπη δίνει λύσεις και βοηθάει την ευμαριά τους ενώ μερικές φορές ο κόσμος μπορεί να πιστεύει το αντίθετο. Αυτό είναι αδικαιολόγητο αλλά είναι μια πραγματικότητα. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο Αλένα Μασούρ. Ε- ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου για την παρουσία του Μισελ Σαπά εδώ. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε σε πολλά θέματα στον τομέα της φορολογίας, της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Οι θέσεις της γαλλικής κυβέρνησης είναι σωστές. Σε τομείς όπως οι νέοι ήδη πόροι, η φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η βασική φορολογική ε, βάση για τις επιχειρήσεις. Αλλά εδώ και λίγες εβδομάδες μάθαμε από το κρατικό κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης ότι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που ελέγχονται από το κράτος χρησιμοποιούν μαζικά φορολογικές υπεκφυγές θα έλεγα όπως ε, τα αεροδρόμια του Παρισιού και άλλες εταιρείες πώς η γαλλική κυβέρνηση θέλει να είναι αξιόπιστη στη Γαλλία απέναντι στους φορολογουμένους και στην Ευρώπη απέναντι στους εταίρους της, αν οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχει δίνουν το κακό παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ερώτησή σας η οποία είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Κοιτάξτε, εγώ σας απαντώ ειλικρινά. Αυτά τα οποία, στα οποία αναφερθήκατε ισχύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και επειδή ισχύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό εντάσσονται στους μηχανισμούς λειτουργίας και στις διαδικασίες πρόσκλησης κερδών πολλών επιχειρήσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι πιο απαιτητικός από εσά. Το θέμα δεν τίθεται μόνο για τις επιχειρήσεις που ελέγχει άμεσα, το κράτος αλλά και για τις επιχειρήσεις τις οποίες είναι παρόν το κράτος, η Ρενό σαν παράδειγμα. Είμαστε παρόντες σε ένα επίπεδο που μπορούμε να μπλοκάρουμε μία απόφαση αλλά όχι όμως ε, πλειοψηφικά, δεν παίρνουμε εμεί τις αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή το κράτος λοιπόν είναι παρόν σε μια επιχείρηση. Θα πρέπει να απαιτήσει καταρχάς από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης να λειτουργήσει με υποδειγματικό τρόπο. Εγώ έχω απαιτήσει τον υποδειγματικό χαρακτήρα στη συμπεριφορά όλων αυτών των επιχειρήσεων στις οποίες στο Διοικητικό του Συμβούλιο υπάρχει κράτος. Θυγατρικές επιχειρήσεις. Πού είναι οι θυγατρικές επιχειρήσεις, τι νόημα έχουν οι θυγατρικές επιχειρήσεις, διεύρυνση δραστηριοτήτων, αν αυτός είναι ο στόχος, τόσο το καλύτερο. Αν ο στόχος των φυγατρικών σε άλλες χώρες είναι η φοροαποφυγή, όχι βέβαια, θα υπάρξει λοιπόν έλεγχος. Κάποιες από τις επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να δημοσιεύουν τον κατάλογο των φυγατρικών τους. Θα είμαι απόλυτος κάθετος σε αυτό. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ειδικέ βολικές φορολογικές ρυθμίσεις και φυσικά δεν μπορούμε παρά να είμαστε απόλυτα απαιτητικοί απέναντι στις κρατικές επιχειρήσεις. Μαρία Ζωαρντρίγης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εμεί θέλουμε να χαιρετήσουμε την ε, δέσμευση που ανέλαβε η γαλλική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την αναθέρμανση της διαδικασίας συμπλήρωσης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Γνωρίζουμε όμως ότι ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι το θέμα της ανάγκης να υπάρξει μια ειδική ε, ρύθμιση, ένα είδος προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ αποκλειστικά και μόνο. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο η γαλλική κυβέρνηση είναι ανοιχτή για μια τέτοια ιδέα. Τι πιστεύετε σε σχέση με το ρόλο που μπορεί να διαδραματιστεί από ένα τέτοιο προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Μπορεί να βοηθήσει τη διαθροτική σύγκληση, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ε, υποστήριξη στον κοινωνικό τομέα, μπορεί να υποστηρίξει την αντιμετώπιση των ε, ασυμμετρικών κλειδονισμών. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> κυρία Βουλευτά. Και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, γίνονται συζητήσεις σε βάθος και φυσικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εδώ είναι ο πυρήνα τη λειτουργία του ω αρχή του προπολογισμού και υπάρχουν πολλέ συζητήσει που γίνονται στι χώρε μα. Αν σκεφτώ για τις ε, τωρινές συνθήκες, μάλλον αν βγω από τις τωρινές συνθήκες, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει ένας χωριστός προϋπολογισμός με ίδιους πόρους που είναι απαραίτητο για να γίνει για την ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και για την δημοκρατική ε, έκφραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι πάντα η προοπτική προς την οποία κινούμεθα. Σήμερα όμως Έχουμε 11 κράτη-μέλη που επεξεργάζονται την ιδέα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μια δυνατή χρησιμοποίηση αυτού του φόρου θα μπορούσε να, να αποτελέσει ένα ίδιο πόρο, ο οποίος θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρώπη εν γέννη να ακολουθήσει πολιτικές αλληλεγγύης καταρχήν στο έδαφος της αλλά και αλληλεγγύης έναντι άλλων περιοχών του πλανήτη μας προσωπικά υποστηρίζω ιδιαίτερα το να μπορέσει η Ευρώπη να είναι ακόμα πιο παρούσα στην υποστήριξη των αναπτυσσομένων χωρών και ιδίως μέσα στα πλαίσια του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κεφαλαιόδες ζήτημα, ένα θέμα που είναι παγκόσμια σημασία και που είναι ένα θέμα που η Ευρώπη μπορεί να είναι σημαντική και υποδειγματική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη Γαλλία γιατί μέχρι το τέλος του έτους θα υποδεχτεί την COP21, τη διάσκεψη κορυφής για την κλιματική αλλαγή και αυτό σημαίνει ότι είμαστε και απόλυτα διατεθειμένοι να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της COP21, αλλά και γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αποκρισταλώνει την θέληση της Ευρώπης. Έχουμε την ικανότητα σε επίπεδο καινοτομία, σε επίπεδο χρηματοδότησης για να προωθήσουμε σχέδια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν να είναι μια λύση, να επιτρέψουν σε χώρες που έχουν μεγάλες δυσκολίες να προσαρμοστούν στις προκλήσεις αυτές τη κλιματική αλλαγή αλλά και τι οικονομίε μα να προχωρήσουν προ μια μείωση τη κατανάλωση ενέργεια και τη μετρίαση τη αλλαγή του κλίματο. Φυσικά αυτή τη στιγμή έχουμε τους περιορισμούς λόγω του προϋπολογισμού του εθνικού. Κανένας υπουργό προϋπολογισμών οικονομικών δεν θέλει να προκύψουν πρόσθετοι πόροι που θα φύγουν από το θησαυροφυλάκιό του. Αυτό θα δυσκολέψει λοιπόν την κατάσταση του εθνικού προϋπολογισμού. Για να μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε θα πρέπει να περιμένουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα που αναφέρατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ε, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, τον οποίο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του, ε, για να θέσω ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης στο Eurogroup. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, ε, οι οποίες πέρα από, την, το πολιτικό ενδιαφέρον που δημιουργούν, δημιουργούν και προβλήματα στη λειτουργία της οικονομίας. Δηλαδή, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι δεν θα σταθεροποιηθεί το πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας, άλλοι τραβάνε τα λεφτά τους από τις ελληνικές τράπεζες και διάφορα τέτοια. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Τι ακριβώς συζητάτε στο Eurogroup. Συζητάτε την τετράμινη παράταση του υπάρχοντος προγράμματος σύμφωνα με, ε, με βάση τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Συζητάτε κάτι παραπάνω που είναι πολύ πιο σημαντικό, δηλαδή την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου για το 2015 και το 2016 ή ε, γίνονται παράλληλα αυτές οι διαδικασίες, δηλαδή πάτε για την τετράμινη παράταση ενώ προετοιμάζεστε, ενώ ζεσταίνεστε και για, τη για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού το 2000... του 2015 και, το... και του 2016. Θα θέλαμε να τα ξέρουμε αυτά ε, σαν ε, πολιτικοί αλλά κυρίως σαν πολίτες γιατί από την απάντηση ε, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και τις δυνατότητές της να, πρώτα να σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας η οποία αφορά άμεσα τη χώρα σας φυσικά αλλά αφορά και το σύνολο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα πλαίσιο ανάκαμψης οικονομικής της Ευρωζώνης, χαμηλής ανάκαμψης, αλλά έχουμε ανάγκη εμπιστοσύνη. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από την εμπιστοσύνη. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει ανάγκη την εμπιστοσύνη, από την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, η καταστροφή της Ελλάδας οικονομικά δεν θα ήταν ίσως μια καταστροφή οικονομικά της Ευρωζώνης, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο αρνητικό. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε διαρκείς λύσεις για την Ελλάδα. Τι συζητάμε. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι το τρέχον πρόγραμμα. Πρέπει να κλείσει το τρέχον πρόγραμμα. Να δούμε πού βρισκόμαστε, τι εξελίξεις έχουν υπάρξει, ποιες ήταν οι επιθυμητές εξελίξεις, ποιες ήταν οι απαραίτητες αυτές που έχουν σημειωθεί, να δούμε πού βρισκόμαστε και σε σχέση με τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου και με τελική προθεσμία το τέλος του Ιουνίου. Ταυτόχρονα όμως συζητάμε όχι ένα νέο πρόγραμμα, αλλά εξετάζουμε την συνέχεια των πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο ουδέτερο. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα έχει ανάγκη την συνέχεια της συνοδείας της Ευρωζώνης, όχι ίσως με τον ίδιο τρόπο, όχι με τα ίδια ποσά και όχι με τα ίδια μέσα, αλλά έχει ανάγκη συνοδείας περαιτέρω έτσι ώστε η επιστροφή της ανάκαμψης να είναι μια διαρκής επιστροφή έτσι ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να μπορούν να πάρουν μεσοπρόθεσμες αποφάσεις έτσι ώστε οι καταθέτες να βάζουν χρήματα στις τράπεζες και όχι να τα Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να υπάρξει μια αποκατάσταση ενός κλίματος ηρεμίας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να ανακάμψουμε, να επιστρέψουμε στην ανάκαμψη, κάτι που έχει λείψει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ίσως κάτι τέτοιο ήταν αναπόφευκτο στο παρελθόν. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ανάπτυξη. Η κυρία Μπερές έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και για τις γενικές σκέψεις σας, για αυτά τα οποία λέτε, ότι αυτά που κάνετε στη Γαλλία τα κάνετε και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη. Μας είπατε επίσης ότι θα πρέπει να προσέξουμε τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και να πω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και το πού θέλουμε να πάμε από εδώ και πέρα. Πέρα από τις αλλαγές της συνθήκης θα πρέπει να έχουμε μία άποψη για το τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ορίσουμε κάποια στάδια, κάποιες φάσεις. Και εδώ τίθεται το θέμα της δημοσιονομικής εισαγωγικά ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ήδη και είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει ίσως εναρμονισμένα με μια άλλη συζήτηση που θα ξεκινήσει σύντομα σχετικά με τον προϋπολογισμό αυστηρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί το θέμα των ιδίων πόρων. Αν θέλουμε περισσότερες δημοσιονομικές δυνατότητες στην ε, ζώνη ευρώ, τότε φυσικά θα τεθεί επίσης και το θέμα εδώ των ιδίων πόρων της Ευρωζώνης. Με λίγα λόγια, πώς θα χρηματοδοτήσουμε αύριο περισσότερη αλληλεγγύη ανάμεσα στους Ευρωπαίους για να κερδίσουμε και την μάχη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Σήμερα είμαστε σε μια πρώτη φάση με το ε, επενδυτικό πρόγραμμα. Ε, Juncker. Είναι μπροστά μας το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα στην ουσία ε, είναι καλοδεχούμενο, αλλά είναι μικρό αυτό το πρόγραμμα και σε λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το πρόγραμμα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για την Ευρωζώνη, τι μπορούμε να κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω ενός πραγματικά επενδυτικού προϋπολογισμού. Αυτό τίθεται και για την Ευρωζώνη και για τις χώρες της και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάνω σε όλα αυτά πώς βλέπετε την συζήτηση για το γενικότερο θέμα του ιδίου πόρους. Πράγματι είναι μια συζήτηση ουσίας εδώ και είναι φυσικά πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Επαρέχομαι πάντα σε αυτό το σημείο. Σας λέω ότι το πλαίσιο το, του προπολογισμού στις χώρες μας είναι δύσκολο για άλλες μας τις χώρες. Είμαστε σε μια αν ήμασταν σε μια εποχή μεγαλύτερη χαλαρότητα για τον προπολογισμό στι χώρε μα, θα είχαμε μεγαλύτερε δυνατότητε για να εφαρμόσουμε αυτού του ίδιου πόρου και να επικρατήσει περισσότερο μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, ένα ευρωπαϊκό πνεύμα, να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε πολιτικέ, οι οποίε, όπω είπατε πολύ σωστά, είναι πολιτικέ αλληλεγγύη για όλο το ευρωπαϊκό έδαφο. Και επίση αλληλεγγύη σε σχέση με τον κόσμο έξω από την Ευρώπη, με το σύνολο του πλανήτη μα. Το θέμα τώρα των ιδιών Ναι, υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή κάποιες διατάξεις που αφορούν κάποιους πόρους ευρωπαϊκούς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, οι μηχανισμοί που έχουν να κάνουν με την Τραπεζική Ένωση, τα ταμεία επίλυσης και εξυγίανσης των τραπεζών που ουσιαστικά προέρχονται από τις συνεισφορές των τραπεζών. Εδώ έχουμε ήδη κάποιους πόρους αυτού του είδους οι οποίοι έχουν αυτό τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Μπορούμε ήδη να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτούς τους πόρους και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αναπολιτική τέτοιους μηχανισμούς προτού κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα που θα σήμαινε μία αλλαγή στους ίδιους πόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μπορεί να εκφράζεται και η δημοκρατία και η αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο σημερινό πλαίσιο όμως και πάλι αυτή η πραγματιστική άποψη που ανέφερα προηγουμένως είναι αυτή η οποία έχει περισσότερες δυνατότητες να λειτουργήσει. Αλλά ο πραγματισμός δεν είναι ο αντίπαλος της φιλοδοξίας. Ο πραγματισμός είναι χρήσιμο και όταν εγγράφεται σε μια τέτοια προοπτική. Ο κύριος Μουλασάνη. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για κάποια άδικα, κατά κάποιο τρόπο, κλισέ που αναφέρονται σε σχέση με τη Γαλλία και τη γαλλική οικονομία στις αρχικές σας παρατηρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή θα πραγματοποιήσουμε, θα κάνουμε πραγματικό και ένα άλλο κλισέ, ότι οι πολιτικοί μιλάνε με ωραία λόγια, αλλά δεν ακολουθούνται τα λόγια αυτά από πράξεις το να έχουμε ένα κατάλογο μεταρρυθμίσεων για, τις, για τη Γαλλία, αυτός ο κατάλογος είναι πιο μεγάλος, πιο μακρύς από αυτά που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν. Γιατί λοιπόν η Γαλλία έχει τόσες δυσκολίες να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και που άλλες χώρες έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν τα τελευταία χρόνια. Θέτω αυτό το ερώτημα καλή την πίστη γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή και ανταγωνιστική γαλλική οικονομία η οποία είναι κεφαλαιώδης για να έχουμε μια πραγματικά ανταγωνιστική οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο. Και όταν μιλάμε λοιπόν για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανταγωνιστικότητα, η, τα ερωτήματά μου ποια είναι τα σχέδιά σας για να μειωθεί το εργασιακό κόστος, για να μειωθούν οι ακαμψίες στην αγορά εργασία. Γιατί όπω έχουμε δει, η ευκαμψία στι αγορέ εργασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερε επενδύσει. Και το άλλο συγκεκριμένο ερώτημα μου είναι το εξή. Η Γαλλία έχει ένα σχετικά υψηλό κατώτατο μισθό. Μήπω βλέπετε ότι αυτό είναι μία από τι αιτίε για το σχετικά υψηλό επίπεδο ανεργία των νέων στη Γαλλία και αν έχετε σχέδια να πράξετε κάτι σχετικά. Και το τελευταίο μου ερώτημα, ακολουθώντα αυτά που είπε η κυρία η Εστέρ προηγουμένω, όταν μίλησε για το θέμα των ελλημάτων και των πλεονασμάτων μέσα στην περιοχή του ευρώ, είπατε εκεί πέρα ότι πρέπει να έχουμε την ότι αυτό που μετράει είναι η συνολική εικόνα της Ευρωζώνης. Πιστεύετε ότι οι ανισομέρειες μέσα σε μια νομισματική περιοχή, ενιαία περιοχή, δεν έχουν καμία σημασία. Ευχαριστώ. οι οι ελλείψεις ισορροπίας στο εσωτερικό της Οικονομικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει την κατάσταση και πρέπει να καταπολεμηθεί μέσω πολιτικών σύγκλησης, σαν παράδειγμα κοινωνικής σύγκλησης και έρχομαι εδώ στον κατώτατο μισθό. Μπορούμε να μιλήσουμε για το κόστος της εργασίας, μπορούμε να μιλήσουμε για τους μηχανισμούς καθορισμού του κόστους της εργασίας, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπάρξει και μια κάποια κοινωνική σύγκληση. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορές οικονομικές, υπάρχουν διαφορές ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν όμως και κοινωνικές διαφορές. Σεβόμενοι λοιπόν την κάθε χώρα, σεβόμενοι την αγοριστική ικανότητα της κάθε χώρας, σεβόμενοι τα έθιμα κάθε χώρας, βλέπουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο κοινέ ρυθμίσεις ο κατώτατος μισθός σαν παράδειγμα σε ορισμένες χώρες είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου, σε άλλες χώρες είναι απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν και εδώ πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Είπατε με καλή πρόθεση γιατί είναι τόσο δύσκολο στη Γαλλία να μεταρρυθμιστεί. Ε, γιατί είναι τόσο δύσκολο για την Γαλλία να πείσει ότι μεταρρυθμίζεται, ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις. Μήπως είμαστε φυλακισμένοι μιας εξωτερικής εικόνας. Δύο παραδείγματα. Λέτε γιατί δεν μειώνεται το κόστος της εργασίας. Ε, αυτό δεν κάνουμε. 40 δις μείωση σε τέσσερα χρόνια. Αυτό επέτρεψε φέτος να ανέβουν σιγά σιγά οι επιχειρήσεις. Και αυτό επιτρέπει στις γαλλικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να επενδύσουν το 2015 αύξηση των επενδύσεων 7%. Μεταρρυθμιζόμεθα λοιπόν. Ίσως να μην φαίνεται εύκολο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά οι αλλαγές έρχονται. Η καλή σας θέληση λοιπόν πρέπει να γίνει πιο εφαρμοσμένη λίγο για να δείτε τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται και τις μεταρρυθμίσεις που, που ξεκινάνε. Για την αγορά εργασίας. Εμείς μεταρρυθμίσαμε αυτό που ονομάζουμε συλλογικές απολύσεις, άνω των 11 υπαλλήλων για οικονομικούς λόγους. Δεν μιλάω για μεμονωμένες επιχειρήσεις. Μια εταιρεία δεν πάει καλά, ένα εργοστάσιο δεν πάει καλά. Πρέπει να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων. Πώς το κάνει αυτό. Η ρύθμιση στη Γαλλία πάντα ήταν πολύ δύσκολη υποτίθεται, κόστιζε πολύ και ήταν αβέβαιη. Τώρα δεν ισχύει αυτό, έχει αλλάξει εντελώς. Και έχει αλλάξει μετά και από συμφωνία με τα συνδικάτα και την εργοδοσία. Αυτή δεν είναι η εικόνα που δίνει η Γαλλία συνήθως. Παρόλα αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κατάσταση των Γκουντιέρ σαν παράδειγμα που έγινε γνωστή στον κόσμο. Γιατί πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μια σύγκρουση. Υπήρχε αβεβαιότητα για την επιχείρηση και για τους εργαζομένους. Αυτό δεν επαναλαμβάνεται πια στη Γαλλία γιατί έγινε η μεταρρύθμιση. Πρέπει να την γνωστοποιήσουμε ίσως, πρέπει να την κατανοήσετε. Πρέπει να συνεχίσουμε τις αλλαγές φυσικά. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αναγνωρίσετε ότι η Γαλλία είναι ικανή να κάνει μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη και κυρίως πολύ επικοδομητική η επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους. Uh, Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ε, και σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου δεν, ε, δεν απαγορεύεται από τις συνθήκες, θα ήταν προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ που μας το θυμήσατε. Πάντως Νομίζω ότι τα τελευταία στοιχεία πράγματι δείχνουν ότι ακολουθούμε τον σωστό δρόμο, ένα δρόμο ανάκαμψης. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, διακυβέρνησή μας την οικονομική. Ακούστηκαν απόψεις, συζητήθηκαν απόψεις, χρήσιμες απόψεις για το μέλλον. Λοιπόν θα συνεχίσουμε τον διάλογο μαζί σας, θα συνεχίσουμε τον διάλογο με τη χώρα σας και σας ευχαριστώ που πήρατε μέρος στις συζητήσεις μας έτσι ώστε να έχουμε μια φιλόδοξη και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. 26 Μαΐου η επόμενη συνάντηση, τρίτη απογευματινή. Τέλος.